Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε να ψηφίσουμε Καθίστε όμως παρακαλώ. Wir haben zur Abstimmung lediglich die Entschließung. Έχουμε να ψηφίσουμε την απόφαση για το άνοιγμα των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων σε σχέση με το σύστημα αρρωγής για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα σχολικά ιδρύματα. Ξεκινούμε με κάποιες τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας Unblock. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά. Θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία έλεγχου. Ψηφίσατε όλοι όλες. Κάποιοι συνάδελφοι τρέχουν ακόμα. Φαίνεται ότι έχουν ψηφίσει όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά α... Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία ελέγχου για την τροπολογία 30. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 θέλετε έλεγχο για την 37 μάλιστα αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 19. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 50 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. <clears throat> Η 22 εκπίπτει λοιπόν. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 έλεγχος για την 28 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία έλεγχου Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 66. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2 και 53 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές <clears throat> θα πρέπει να ελέγξουμε. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε πράγματι. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τεκτή. Η 56 εκπίπτει ως εκ τούτου. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει 58. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει 59. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκπίπτει το αρχικό κείμενο τροπολογία 57 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται εκπίπτει 63 ως εκ τούτου. Συνολική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε πληροφορίε Εγκρίθηκε. Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτω μέχρι τις 7 την Σύνοδο Λομέλειας.